Αρχίζουμε λοιπόν με τη συνάντηση αυτή του απογεύματο. Πρόκειται για το διορισμό μέλους του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανση. Καλωσορίζω εδώ τον Πέδρο Ματσάδο που προτείνεται ω υποψήφιο για μέλος του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκρόασή μα βασίζεται στο άρθρο 56 του κανονισμού του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανση που λέει ότι το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση για ορισμό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των ε, πλήρων μελών ε, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης μετά από έγκριση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Κοινοβούλιο. Βάσει λοιπόν ε, των πρακτικών που έχουν συμφωνηθεί θα ακούσουμε πρώτα για 5 λεπτά τον κύριο Πέντρο Ματσάδο και μετά τέσσερα λεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις με επερώτηση εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος. Κάθε πολιτική ομάδα θα έχει μια περίοδο στη διάθεσή του και αν το επιτρέψει ο χρόνος θα έχουμε επιπλέον δύο λεπτά στη διαδικασία Catch the Eye για τον κάθε ερωτούντα ακολουθώντας τη σταθμισμένη προσέγγιση βάσει πολιτικών ομάδων. Εάν ο χρόνος επίσης επιτρέπει και εφόσον το επιθυμεί ο κύριος Ματσάδο θα μπορέσει να κλείσει με δύο λεπτά παρέμβαση στο τέλος. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Πέντρο Ματσάδο τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Αγαπητοί Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, είναι τιμή και μεγάλη ευθύνη για μένα που έρχομαι εδώ στην ακρόαση αυτή βάσει της υποψηφιότητά μου για μέλος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης. Η διαφάνεια και λογοδοσία με ενώπιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατική νομιμότητα. Θα αρχίσω παρουσιάζοντας τις απόψεις μου για το θέμα της εξυγένσης. Θα σας μιλήσω για την επαγγελματική μου εμπειρία, τη σταδιοδρομία μου και γιατί θέλω να αναλάβω αυτή τη θέση. Υπάρχει το ενίο Συμβούλιο Εξυγένσης και ο σχετικός μηχανισμός που αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα στην ε, οικοδόμηση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Δεν ε, θα πρέπει να μην υπάρχει εξυγίανση στους πυλώνες της εξυγίανσης. Το νέο Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει φροντίσει να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες με την οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών αλλά και για τον νέο μηχανισμό. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε καλό επίπεδο λειτουργίας, πλήρους λειτουργίας, με σχεδιασμό και με τους στόχους για το ημερέλ πρόσφατα. Αλλά η εξυγίανση δεν λειτουργεί μέσα σε ένα κενό. Απαιτείται ένα ε, πλαίσιο νομοθετικό. Θα σας αναφέρω κάποιες προκλήσεις που πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας. Πρώτον, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Οι περισσότερες τραπεζικές ομάδες είναι υπό τη δικιά μας εποπτεία, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Οι διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά την ομοθεσία στις χώρες μέλη για την ε, εξυγίανση των τραπεζών ή για την ρευστοποίησή τους είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Και έτσι λοιπόν πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε την, ε, τις συνταγματικές προϋποθέσεις τουλάχιστον στο πλαίσιο της ευθοποίησης των τραπεζών, χρειάζεται κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, κάτι που απορρέει από το πρώτο, ο ρόλος του προγράμματος για την εγγύηση καταθέσεων. Όσοι δεν, όσες τράπεζες δεν καταφέρουν να περάσουν τις δοκιμασίες, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τον μηχανισμό εγγύησης. Μπορούμε λοιπόν να επωφεληθούμε από την εμπειρία που έχουμε συλλέξει σε άλλες δικαιοδοσίες. Επίσης, η εξυγίανση θα πρέπει να υλοποιείται αποτελεσματικά. Αμέσως μετά την εξυγίανση θα πρέπει να προχωράμε στα επόμενα στέδια ώστε να υπάρχει πάντα η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Μπορεί να υπάρχουν ε, λοιπόν ε, δίκτυα προστασίας και για να είμαστε σίγουροι το backstop του Συμβουλίου Εξυγένσης φροντίζει για την ρευστότητα που χρειάζεται. Η διευκόλυνση αυτή αποτελεί και το βασικό στοιχείο της εξυγένσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στην εξυγένση συνολικά. Έπειτα, το πλαίσιο του MRL έχει να κάνει με την απορρόφηση. Η πολιτική του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης έχει να κάνει με τις ομάδες εκείνες τραπεζών που δεν είναι σε θέση να μπορούν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην αγορές. Και αυτό συνοδεύεται και με την δυνατότητα εξυγένσης. Επίσης, το θέμα των ε, απρόπτων στην εξυγένση. Εγγύησεις τρίτων νομερών άλλες εγγύησεις και ιδιαίτερα οι επίμαχες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την αποτελεσματικότητα του δεύτερου πυλώνα και δεν αποκλείει ο νόμος τέτοια εξυγίανση. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε τι έχουν οι ισολογισμοί των τραπεζών. Εδώ έχουν να κάνουν νομοθετικές διαδικασίες που ισχύουν στην κάθε χώρα που μπορεί να επηρεάσουν τις ανάγκες κεφαλοποίησης και υπάρχει και ανάγκη να μαθαίνουμε από τις εθνικές αρχές και τις δικές τους εμπειρίες από το παρελθόν, ώστε να προβλέψουμε τις εξελίξεις. Το νέο πλαίσιο εξυγένσης δεν υπάρχει μόνο με νομοθετικές ε, πράξεις, αλλά είναι και ένας ζωντανό οργανισμός, Οπότε χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στο νέο Συμβούλιο Εξυγένσης και τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές. Τώρα, έχω επαγγελματική εμπειρία που με κάνει να πιστεύω ότι είμαι κατάλληλος για το διορισμό αυτόν. Από το 2001 έχω ειδικευτεί στην ομοθεσία για την εξυγένση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω αναλάβει διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες που κατέληξαν σε ενδιαφέροντα προγράμματα μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Από το 2001, λοιπόν, έχω αναλάβει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εποπτεία και πρόσφατα και για την εξυγένση. Δίνω μεγάλη σημασία στην εξυγένση γιατί αποτελεί μέρος του έργου μου σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας μου τα τελευταία δέκα χρόνια. Συντόνισα, ε, για παράδειγμα, ε, στο πλαίσιο εξυγένσης στην Πορτογαλία, στην αρχή της κρίσης. Μετά Ήμουνα στην τράπεζα της Πορτογαλίας, στην Κεντρική Τράπεζα και τους κανόνες που βοήθησαν να διαμορφωθούν τους εφάρμοσα στη συνέχεια και ήδη εφαρμόζονται εκεί στις πιο σημαντικές τράπεζες. Είχα επίσης την ευκαιρία να βοηθήσω τις αρχές της Αντόρας για να εξηγιάνουν μία από τις μεγαλύτερες τραπεζές τους μετά από ένα, ένα μεγάλο σκάνδαλο που είχε να κάνει με το ξέπλυμα χρήματος. Έπειτα υπάρχουν διάφορες επίμαχες ε, περιπτώσεις για άλλες τράπεζες και κάθε φορά με επιτυχή αποτελέσματα προκειμένου να προχωρήσει το σύστημα εξυγένσης στην Ευρώπη. Έχω μεγάλη εμπειρία λοιπόν με πολλές προκλήσεις που έχω αντιμετωπίσει και έτσι έχω καταλάβει καλύτερα ε, ποια είναι η προσέγγιση και οι διαδικασίες για τη διάσωση μιας ε, τράπεζας, ε, ποιοι επιμερίζονται τις ευθύνες και το κόστος. Βέβαια, πρέπει να διασφαλίζονται όλα αυτά από σωστό σχεδιασμό και από ένα στέρεο πλαίσιο. Η σταδιοδρομία μου με βοήθησε πολύ, αποτελεί ένα δώρο για μένα. Με γνώση σε διάφορους τομείς. Είναι βέβαια μια διαδικασία ε, βάσει της οποίας μαθαίνουμε συνεχώς και πιστεύω ότι και ο ιδιωτικό τομέας μπορεί να βοηθήσει. Από όπου πέρασα κάτι το οποίο με βοηθάει ακόμα περισσότερο στις γνώσεις μου. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετήσω στο νέο Συμβούλιο Εξυγίανσης και να βοηθήσω την Τραπεζική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα γενικότερα. Thank you very much. Now we move on. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στον Μάρκους Φέρμπερ του ΕΛΚ για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστούμε κύριε Ματσάντο και καλώς ορίσατε. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εξυγίανση. Καταλαβαίνετε γερμανικά τέλεια για την εξηγένση των τραπεζών είναι η σωστή αξιολόγηση του ενεργητικού. Ειδικότερα όταν αυτά είναι χαμηλότερης αξίας. Συνήθως στην εξηγένση υπάρχει πίεση χρόνου και το κριτήριο για τους πιστωτές ή όχι δεν είναι εύκολο. Στην Banca Popular τότε το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αμφισβήτησε πολλά πράγματα και απέτησε κάποιες εκθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τι συμπεράσματα ε, έχετε αποκομίσει για την δουλειά του Ενίου Ταμείου Συμβουλίου Εξυγένσης. Το πλαίσιο που έχουμε ε, δημιουργήσει είναι αυτό το οποίο θα ε, κρίνει αν θα είναι αποφασιστικός ο μηχανισμός αυτός. Τώρα, για να κάνει κανείς αυτό ε, την εξυγένση θα πρέπει πριν προχωρήσει ε, να έχει γίνει μια αξιολόγηση και της μεθοδολογίας που θα ακολουθεί για την εξυγένση και η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να βασίζεται όπως και η αξιολόγηση σε στέρεα κριτήρια τα οποία σχετίζονται με τη σχέση με την ε, προληπτική προσαρμογή στην δίκαιη αξία. Είναι δηλαδή τα κριτήρια τα οποία ουσιαστικά οδηγούν σε μία ε, αξιολόγηση ε, κοντά στην αξία αγοράς και όχι σε μία ε, αξία η οποία θα προσεγγίζει την έννοια του ξεπουλήματος. Οπότε αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, για την αξιολόγηση την ίδια, αυτό το οποίο θα πρέπει να ορίζουμε και έτσι το καταλαβαίνω γιατί νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ε, στο ενίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, είναι ότι δημιουργούμε το πλαίσιο για την στέρεη αξιολόγηση ε, με το ε, Σαββατοκύριακο που πάντα είναι ο χρόνο που έχουμε για να, να προετοιμάσουμε μαζί την αξιολόγηση. Οπότε όταν ξανανοίξει Δευτέρα το πρωί η τράπεζα, άσχετα με την εξυγίανση που θα γίνει, έχουμε μία πλήρη απορρόφηση της ζημίας αυτό είναι ο πιο στέρος τρόπος για να προχωρήσει κανείς. Αλλά ε, είναι ουσιαστικά και ο τρόπος για να εξασφαλίσουμε πως μετά η επανακεφαλαιοποίηση θα γίνει και αυτή σε στέρεη και σωστή βάση. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το πιο ουσιαστικό για να εξασφαλίσουμε πως η αξιολόγηση ε, της τράπεζας θα είναι η σωστή. Τώρα, με αυτό σχετίζεται ένα πρόβλημα με το οποίο πολλές φορές έχουμε προβλήματα. Και αυτό είναι και ε, ε, το πρόβλημα που είχα με την εκαθάριση της τράπεζας του Σάντου. Ξεκινάμε με τον ισολογισμό ως, πριν την εξυγίανση. Ως είχε. Και ίσως εκεί δεν είναι γραμμική η προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο για να δούμε ποιες θα είναι οι απαραίτητες προσαρμογές που πρέπει να κάνουμε πριν την εξυγίανση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των δύο ημερών κάνουμε μια ερμηνεία της αξιολόγησης και πολλές φορές δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ή έτοιμοι να στήσουμε μία στέρεη προσαρμογή η οποία θα απηχεί πλήρως όχι μόνο την απορρόφηση της ζημίας και το ποσό που χρειάζεται, αλλά παράλληλα και το ποσό που χρειάζεται για την επανακεφαλαιοποίηση. Οπότε, τότε, για να διορθώσουμε αυτή την ε, έλλειψη ε, ορθής αξιολόγησης, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε συνέχεια ε, τις διακυμάνσεις στην αξία των περιουσιακών στοιχείων ή της τιμής ε, είτε στον ισολογισμό που προκύπτει ε, μετά το Σαββατοκύριακο εξυγίανσης είτε μετά αφού ξεκινήσει αυτή. Είναι λοιπόν ουσιαστικά πολύ κρίσιμο η προσέγγιση για την αξιολόγηση που έγινε το Σαββατοκύριακο να είναι η σωστή. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι έτοιμοι να συνεχίσουμε να κάνουμε τις προσαρμογές, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η αξιολόγηση θεωρείται τελεσμένη Γιατί μόνο αυτό θα δώσει σιγουριά στην αγορά. Και αυτό δείχνει η εμπειρία μας. Ότι μετά από κάποιες εβδομάδες με την τράπεζα του Σάντου καταφέραμε να κλείσουμε ε, τον ε, ε, αρχικό προσωρινό ισολογισμό και να τον κλείσουμε με κάποιες προληπτικές προσαρμογές έτσι ώστε η τράπεζα να μπορέσει να συνεχίσει και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Τώρα, για να κλείσω στα γρήγορα τούτο. Δεν σχετίζεται με μία από τις υποθέσεις που θα θέσετε εσείς, που ε, είναι το, η Banco Popular. Αυτή ήταν ε, μια άλλη αξιολόγηση που γίνεται διαφορετικά και ανεξάρτητα, οπότε ουσιαστικά τίθεται σε κατάσταση χρεοκοπίας και εξετάζει εσύ την αξιολόγηση από πλευράς πιστωτών. Με παραδοχή ότι, ή θα γίνει, ε, ότι θα γίνουν δύο σενάρια συγκρίσιμα μεταξύ τους, ένα εξυγίανσης και ένα εκαθάρισης. Οπότε οι μέτοχοι μπαίνουν σε μία ε, κατηγορία όπου ε, δεν ε, την χάνουν της ίδιας ευνοϊκής αντιμετώπισης όπως σε μία περίπτωση, περίπτωση γιατί κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την έκθεση που έχουν. Ο κύριος Περέιρα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Ματσάδο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επαγγελματική σας πορεία και η μεγάλη σας ε, εμπειρία στον τομέα της ρύθμισης των τραπεζών και της εποπτείας των τραπεζών του χρηματοπιστικού συστήματος, όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά και στην Ευρώπη. Αυτή η εμπειρία και τα εξαιρετικά σας ε, προσόντα ως νομικού είναι πτυχές που διασφαλίζουν ότι είστε ο κατάλληλος υποψηφίος. Ωστόσο θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσάς τι γνώμη έχετε για την ευρωπαϊκή εμπειρία όσον αφορά την εξήγηση των τραπεζών. Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι κανόνες της εξήγησης των τραπεζών, δεδομένων και των τελευταίων εξελίξεων, ε, ε, μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω ή αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πτυχές που χρειάζονται διόρθωση όσον αφορά για παράδειγμα την αξιολόγηση και από την εμπειρία που έχετε στην Πορτογαλία με την εξυγίανση της τράπεζας Σπίριτου Σάντου ε, θα έχετε αποκτήσει κάποια εμπειρία στην Πορτογαλία που πολύ ειλικρινά ήταν μάλλον τραυματική από πολλές πτυχές. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που εδώ ε, χρησιμοποιήθηκε αυτό το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήθελα να μου πείτε Κατά την άποψή σας, από τα λάθη του παρελθόντος, τι θα πρέπει να μάθουμε, κυρίως ε, από αυτή την υπόθεση συγκεκριμένα και το κανονιστικό πλαίσιο, τι μορφή θα πρέπει να έχει, ούτως ώστε αυτή η εξυγίανση να αντιστοιχεί και στις ανάγκες εξασφάλισης της σταθερότητας ε, της ε, χρηματοοικονομικής αγοράς. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα ε, λειτουργικά ε, να σας πω πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε και μετά να δούμε το ευρύτερη εικόνα όσον αφορά το ε, πλαίσιο εξυγίανσης. Το κλειδί για την εξυγίανση μιας τράπεζας είναι να διατηρείς την ευελιξία στον σχεδιασμό της εξυγίανσης. Μπορεί η ιδιαίτερη περίπτωση ε, ε, μια συγκεκριμένη τράπεζα όσον αφορά την εξηγένση να μην είναι αυτή που έχει ακριβώ προβλέψει στο σχεδιασμό τη εξηγένση. Οπότε απαιτείται κάποια ευελιξία και κάποιε πρόσφατε υποθέσει το αποδεικνύουν ότι δεν κάνει πάντα αυτό που έχει σχεδιάσει, διότι υπάρχουν ιδιαιτερότητε που σε κάνουν ε, στην περίπτωση μια συγκεκριμένη εξηγένση μια συγκεκριμένη τράπεζα να υιοθετήσει ένα άλλο σύστημα εξηγένση. Ωστόσο, κάτι που κάνει εντύπωση είναι ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εξηγένσης πρέπει να έχεις ε, μια πολύ ακριβή εικόνα για το παθητικό μιας τράπεζας. Αυτό είναι πρώτη της σημασίας για να επιτύχει η εξηγένση. Όσα αρχή εξηγένσης, εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε στα χέρια μας ε, αξιόπιστα δεδομένα όσον αφορά το παθητικό, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά η εξηγένση. Ειδικότερα μια εξηγένση που βασίζεται σε Μπεϊλίν. Ένα μάθημα που έχουμε μάθει από τον ΠΕΡΣ είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε επίσης ποιο κομμάτι του παθητικού μιας τράπεζας ή, του παθητικού, ή αυτού που έχει ορίσει η τράπεζα ως παθητικό, δηλαδή χρέη τρίτων μερών, όχι παθητικό της ίδιας τράπεζας, αλλά τρίτων μερών, έχει ε, το εκτεθεί σε επενδυτές, λιανικούς επενδυτές. Αυτοί μπορεί να χαρακτηρίσουν τη φρεγγιότητα μιας τράπεζας ουσιαστικά. Γιατί? Διότι οι λιανικοί επενδυτές ε, τείνουν να είναι και καταθέτες. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν πρόκειται κάποιος ε, να διαγράψει τη θέση το πίστοση ενός λιανικού επενδυτή, αυτό είναι πολύ πιθανό να κινητοποιήσει μια αντίστοιχη συμπεριφορά αυτού και ως καταθέτη, δηλαδή να αποσύρει τις καταθέσεις του γιατί χάνει την εμπιστοσύνη του. Το δεύτερο είναι οι διαφορές, η δημιουργία διαφορών ε, και αυτές ε, ε, προστίθενται στους λιανικούς επενδυτές και αυτό υπονομεύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τώρα Όσον αφορά την ε, κατάσταση αυτή του MRL, να δούμε κατά πόσο ε, ε, χρειάζεται υψηλότερο κατόφλιο για τους λιανικούς επενδυτές, ούτως ώστε αυτοί να έχουν πρόσβαση, να μπορούν να αγοράσουν τέτοιου είδους μέσα. Τώρα, για την ευρύτερη εικόνα θα έλεγα ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργικότητα τη εξυγίανση. Αυτό οφείλεται στην αναντιστοιχεία που υπάρχει μεταξύ του ενιαίου ε, πλαισίου εξυγίανση και των διαφόρων ε, νόμων περιφερειακότητα σε κάθε χώρα, όπου υπάρχουν διαφορετικά σημεία όπου ξεκινάει η εξυγίανση, ε, κάτι που βασίζεται στην αξιολόγηση της αρχής εξυγίανσης. και στο πτωχευτικό δίκαιο της κάθε χώρας αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο ε, μπορεί να επιτρέπει να μην γίνει ε, καθάριση. Οπότε όλα βασίζονται στην αποτελεσματικότητα του πλαισίου εξυγένσης. Ευχαριστούμε πολύ. Λουίς Γκαρικάνο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό το τελευταίο που λέτε για την εξυγένση. Κατά την άποψή σας, η εξυγένση είναι για τους πολλούς ή για τους λίγους. Δηλαδή, αυτοί που έφτιαξαν την οδηγία, την ερμήνευσαν και ήμουνα κι εγώ μεταξύ αυτών, πίστευαν ότι εξυγίανση είναι αν δεν θα γίνει κάτι άλλο. Γιατί πολλοί δεν το θέλουν. Δεν θέλουν ε, την ε, εξυγίανση των άλλων, αλλά θέλουν την εξυγίανση όταν πρόκειται για τη δικιά τους χώρα. Οπότε, αν είναι για τους πολλούς η εξυγίανση, ποιο είναι το ο κλειδί. Πότε κάνουμε εξυγένση και μήπως θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε ότι την εξυγένση την κάνουμε από ένα ή άλλο σημείο, αλλά να είναι το ίδιο για όλες τις χώρες, να υπάρξει εδώ πέρα κάποια εναρμόνιση. Πιστεύετε ότι το πλαίσιο πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή πιστεύετε ότι το ίδιο το πλαίσιο είναι εντάξει ως έχει για το πότε έχουμε εξυγένση και πότε δεν έχουμε. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ βασική η ερώτησή σας για το ίδιο το καθεστώς της εξυγένσης. Εγώ θα προτιμούσα να μην το δω από την οπτική γωνία την ποσοτική, δηλαδή αν είναι για τους πολλούς ή για τους λίγους. Το πλαίσιο της εξυγένσης που έχουμε λέει ότι η εκαθάριση, η πτώχευση ε, γίνεται αν δεν μπορεί ε, να γίνει κάτι άλλο. Αν ε, δεν τηρούνται τα κριτήρια, τότε, για την πτώχευση δηλαδή, τότε πάμε στην εξυγένση ώστε να υπάρχει η σταθερότητα, η οικονομική λειτουργία, η προστασία των καταθετών κλπ. Αυτό που νομίζω πρέπει να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε σε τι βαθμό μία τράπεζα που από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρει, θα πτωχεύσει, κατά πόσο περνάει το κριτήριο του κοινού συμφέροντος. Τι λειτουργίες κρίσιμες εξυπηρετεί αυτή η τράπεζα στις χώρες μέλη και κατά πόσο η οικονομική σταθερότητα θα συνεχιζόταν ακόμα και αν δεν περνούσε στην σε αυτή η τράπεζα, αλλά την αφήναμε να πτωχεύσει. Ίσως να θεωρούμε ότι περισσότερες από τις τράπεζες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι υπόθεση αυτή, ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν τηρούν τα κριτήρια. Το ζήτημα όμως είναι σε τι βαθμό η εκαθάριση σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι αποτελεσματική. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Και ίσως να δούμε ότι έχουμε τέτοια ποικιλομορφία στην ομοθεσία που αφορά την εκαθάριση στις διάφορες χώρες μέλη και όχι μόνο για το τι είναι αυτό ε, το οποίο δημιουργεί, αποτελεί το σημείο κίνησης της όλης διαδικασίας. Πρέπει να καταλάβουμε κατά πόσο θέλουμε την εναρμόνιση όχι, ανάλογα με τη φύση της εκαθάρισης. Τότε θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της εκαθάρισης, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Αν δεν είναι ρεαλιστικό αυτό, τότε, όπως είπα και στην αρχή, στην παρουσίασή μου, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να προσπαθούμε να έχουμε κάποια εναρμόνιση σε αυτό το οποίο βάζει σε κίνηση την όλη διαδικασία. Και μετά να σκεφτούμε και τρόπους ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η εκαθάριση μέσα από ένα καθεστώς όπου θα υπάρξουν και μέτρα στήριξης. υπάρχει το πρόβλημα της μεσαίας τάξης, όπως έχει ονομαστεί και μπορεί να παραμείνει στην Ένωση. όπου τελικά ένας από τους πιο αποτελεσματικούς δρόμους να είναι η εκαθάριση. αλλά συντεταγμένα να αποχωρήσουν από την αγορά μεταφέροντας τα περιουσιακά του στοιχεία ή να στηριχτούν από τα GGS. Ευχαριστώ πολύ. Ορτασούν από τους πράσινους. Ευχαριστώ. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Καταρχήν για το δημόσιο συμφέρον και την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου. Θεωρείτε πως αυτή τη στιγμή είναι ε, αρκετό το νομικό πλαίσιο γιατί είδαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ περιθώριο ε, ερμηνείας του κριτηρίου αυτού. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο αυστηρή η νομική μας προσέγγιση στο πώς αυτό ερμηνεύεται. Δεύτερον, ε, για τα σχέδια εξυγίανσης στο παρελθόν, αυτό που είδαμε είναι ότι καθυστερούμε πάρα πολύ στην προετοιμασία του σχεδίου εξυγίανσης. Εσείς τι σκέφτεστε πώς θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία καλύτερα. Τρίτον, τι γίνεται στην περίπτωση εξυγίανσης όπου έχουμε ε, πιστωτές οι οποίοι έχουν τύχει κακής διαχείρισης. Υπάρχει μηχανισμός που να μπορεί να τους εξασφαλίσει και να τους αποζημιώσει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για το δημόσιο συμφέρον και την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου. Έχετε δίκιο. Είναι ε, μια σαφής έννοια, αόριστη έννοια, η οποία πολλές φορές είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ή ποσοτικοποιούνται και χαρακτηρίζονται με τρόπους που δεν είναι ενδεδειγμένοι. του λεχθέντος. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση του κριτηρίου του δημοσίου συμφέροντος προς εξυγίανση αν ας πούμε αυτή η αξιολόγηση του δημοσίου συμφέροντος δεν είναι απόλυτα αντίστοιχη με αυτή που θα γινόταν στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αξιολόγηση και να πούμε όχι εξυγίανση αλλά ενίσχυση. Ε, ο μηχανισμός για τη διαχείριση τέτοιου κρίσεων στην Ευρώπη θα πρέπει να το δει και πιστεύω ότι εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών ενιών και να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το κριτήριο του δημοσίου συμφέροντος. Ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε νομικά μιλώντας πιο αυστηροί στο πώς το χρησιμοποιούμε. Εγώ προτείνω αυτή τη μεθοδολογία η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πιο αποτελεσματική δεδομένης εμπειρίας που έχουμε ε, αποκτήσει από το παρελθόν. Για τα σχέδια εξυγένσης. Δεν νομίζω ότι πάμε πολύ αργά. Νομίζω ότι είχαμε διάφοροι κύκλοι ε, προγραμματισμού σχεδίων εξυγίανσης από την ε, κίνηση ε, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Σήμερα οι όμιλοι που είναι υπό την αιγίδα μας καλύπτονται πλήρως με τέτοιου είδους σχέδια εξυγίανσης. Αλλά ο κύκλος προγραμματισμού που ξεκινά φέτος, που είναι ο πρώτος ετήσιος για όλους, θα καλύπτει καλύτερα τις βασικές αλλαγές, κυρίως με το MRL, που είναι κομμάτι του πρόσφατου τραπεζικού πακέτου. Δεν θεωρώ πως απαραίτητα, απαραίτητα πως καθυστερούμε. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, για τις τράπεζες που είναι ε, υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Εξυγίανσης, εδώ προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη την διαφορετικότητα των τραπεζικών ομήλων που έχουμε στην Ευρώπη. Γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι τραπεζικές δομές, οι οποίες δεν είναι εύκολο πάντα ε, να περιγραφούν μέσα σε ένα σχέδιο, σχέδιο εξυγένσης. Κάποιες είναι συνεταιριστικές, κάποιες είναι πιο χαλαρά ε, συνδεδεμένες μέσα στον όμιλο, είναι διαφορετικές, επαναλαμβάνω, οι δομές και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως εκεί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κάνουμε μια πραγματική εξυγίανση κανονική και πολλές φορές είναι και οι εθνικές αρχές που οι οποίες δεν έχουν πάντα του απαραίτητου πόρου για να το κάνουν. Οπότε δεν θεωρώ πω εμεί καθυστερούμε. Θεωρούμε, θεωρώ πως ο κύκλος που ξεκινά τώρα είναι πολύ σημαντικός από τον Απρίλιο και μετά. Τώρα, για την κακοδιαχείριση, οποιοδήποτε πιστωτής ο οποίος αποδεικνύει πως έχει τύχει τέτοιου είδους ε, ε, κακοδιαχείρισης θα πρέπει να αποζημιώνεται. Αυτό είναι μια βασική αρχή και αποδεικνύει η εμπειρία μας από την Πορτογαλία. Είναι ουσιαστικό για να διατηρήσει κάποιο τραπεζικό ίδρυμα την άδεια λειτουργίας. Ο κύριος Γκουσμά από την ΚΟΕ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επιστρέψουμε στο ερώτημα της διαδικασίας εξυγίανσης και τους κανόνες στους οποίους βασίζεται αυτή η εξυγίανση. και από την Κομισιόν αλλά και από την Αρχή Εξυγίανσης ακολουθείται μια διαδικασία που συνίσταται στο ότι κάθε διαδικασία εξυγίανσης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό. Διότι αν δούμε τις ε, επιμέρους υποθέσεις ε, εξυγίανσης που είναι συγκρίσιμες και δεν είναι ίδιες, ε, η Κομισιόν, ε, ωστόσο και οι αρχή εξηγενσής όχι μόνο ακολουθούν εντελώς διαφορετικές ε, διαδικασίες, για, για παράδειγμα στην πορτογαλική περίπτωση, ήταν υπερβολική η παρέμβαση. Δεν ήταν η αρχή η ρυθμιστική ουσιαστικά, αλλά η Κομισιόν που υποστήριξε ιδιαίτερα έναν από τους αγοραστές της τράπεζας και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε την αυθαιρεσία εδώ πέρα, αυτή την αυθαιρεσία που εξακολουθεί να υπάρχει, κυρίως όταν η Κομισιόν, η αρχή, η ρυθμιστική αρχή ε, ασκούν τέτοια αυθαιρεσία και όταν ε, ε, τα χρήματα που πρέπει να δοθούν πληρώνονται από τον φορολογούμενο και τότε αυτό που κάνει η αρχή, η ρυθμιστική και η Κομισιόν επηρεάζει μεν και την τράπεζα, αλλά το πληρώνει και ο φορολογούμενο κάθε χώρα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ίδιο να επιρροέσει τι γίνεται μέσα στην ίδια του χώρα, ο φορολογούμενο. Και επίση θέλω να μιλήσουμε για την οικονομική ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από πλευρά ε, Κοινοβουλίου, Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράστηκε η ανησυχία ότι αυτό το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα είναι υπερβολικά κατακρεματισμένο και πρότειναν διάφορους τρόπους για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό του κατακαιρματισμού. Ωστόσο, ο κατακαιρματισμός αυτός είναι που οδήγησε στο ότι πήραμε, φροντίσαμε να μην γίνουν πολύ μεγάλες σε κάποιες τράπεζες. Αν τώρα προχωρήσει η οικονομική ολοκλήρωση, δεν θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε οικονομική συγκέντρωση και σε τράπεζες ε, ε, γίγαντες ε, από τις οποίες θα εξαρτάται το σύστημα. Εγγενώς, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Ε, πολλά τα ζητήματα που αναφέρατε. Το ερώτημα για το πώς κάθε εξηγένση είναι ξεχωριστή περίπτωση. Πριν λίγα λεπτά άκουσα που υπόθηκε ότι πρέπει να διατηρούμε την ευελιξία όσον αφορά την εξηγένση. Θα σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που με το ίδιο εργαλείο εξηγένσης χρειάστηκε ουσιαστικά να επιτύχουμε διαφορετικούς ε, στόχους. Στην περίπτωση της ΜΠΕΣ, αυτό που χρειάστηκε ήταν ένα εργαλείο ε, που μας βοήθησε επειδή δεν υπήρχε αγοραστής. Ε, σε άλλε εξηγιάνσεις έχει αμέσω κάποιον αγοραστή, ο οποίο μπορεί να αγοράσει το κομμάτι τη τράπεζα που παρουσιάζει πρόβλημα. Εκεί δεν είχαμε αγοραστεί. Οπότε για να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα και να διασφαλίσουμε και του καταθέτε, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο γεφύρωση ουσιαστικά. Απλά κάποιο κομμάτι του παθητικού το μεταφέραμε ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη έκθεση για τον ευρύτερο όμιλο ε, ε, και για όλη την ομάδα των καταθών μέσα στην τράπεζα. Στην Banco Espiritu Santo. Στην άλλη περίπτωση υπήρχαν συνέπειε και για τι άλλε περιπτώσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αρχή, αρχέ Ανδόρα έγινε κάτι διαφορετικό. Εκεί θεώρησαν ότι η τράπεζα αποτελούσε κίνδυνο όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Εκεί δημιουργήσαμε μια τράπεζα γέφυρα. Γιατί? Διότι έπρεπε να δούμε τη δέωση επιμέλεια για κάθε. να εφαρμόσουμε. να δούμε τις καταθέσεις, τις κάθε, όλες τις καταθέσεις που υπήρχαν στην τράπεζα και να τις αποδεσμεύουμε ανάλογα με το τι συνέβαινε με αυτές. Οπότε βλέπετε χρησιμοποιούμε το ίδιο εργαλείο γεφύρωσης, απλά προσαρμόζουμε διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε ε, τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και τη διασφάλιση των καταθέσεων και στις δύο περιπτώσεις καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο. Τώρα λέτε ότι φαίνεται να λειτουργούμε κάπως αυθαίρετα ασκώντας αυτές τις εξουσίες. Εγώ θα έλεγα ότι ε, πρέπει να δράση ανάλογα με τη διακριτική ευχέρεια, η οποία διακριτική ευχέρεια θα πρέπει να ε, βασίζεται σε κάποια ε, λογική, σε διάφορες αιτίε. Πρέπει να καταλαβαίνεις γιατί ακολουθείς ένα συγκεκριμένο ε, σύστημα εξυγένσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να συνδυάσεις τους στόχους που προσπαθείς να επιδιώξεις με το μέθοδος εξυγένσης που αποφασίζει να χρησιμοποιήσεις ως αρχή εξυγένσης. Δεν μπορείς νομίζω να μιλάς για ευθερεσία. Ε, έχουμε κάποια διακριτική ευχαίρεια η οποία πρέπει να διατηρείται γιατί είναι θεμελιώδους ε, σημασία και πρέπει να είναι αιτιολογημένη και φυσικά μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ελέγχου. Αλλά για μένα η διατήρηση της ευελιξίας είναι ύψη τη σημασία κατά την εφαρμογή ενό μηχανισμού εξυγένση. Όταν έχει να κάνει με μια ε, ε, τράπεζα που διατρέχει κίνδυνο πτώχευση, ώστε να διασφαλίσει τι καταθέσει και να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα, που για μένα είναι πολύ βασικό, πολύ βασικέ λειτουργίε όσον αφορά την ολοκλήρωση, την οικονομική ολοκλήρωση, τη χρηματοοικονομική, χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα ε, ουσιαστικά είναι ότι έχουμε μια κατακριματισμένη χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη, ειδικότερα μετά από την κρίση. Και αυτός ο καταγραμματισμός δημιουργεί πρόβλημα στην κατανομή των κεφαλαίων. Ε, κάτι που υποχρεώνει τις τράπεζες να δεσμεύουν κεφάλαια ρευστότητα που θα μπορούσαν να διατεθούν στην πραγματική οικονομία. Αν τα πράγματα δεν είχαν έτσι. Εγώ βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι με την εξυγίανση ε, με, συγγνώμη, με την ολοκλήρωση ε, καταλήγει σε τράπεζες γίγαντες. Απλά αντιμετωπίζει ε, την υπερβολική προσφορά που υπάρχει στο σύστημα με αποτέλεσμα ωφέλειες ε, για τους καταθέτες και τους καταναλωτές. Αυτό είναι ο απότερος στόχος της πρόθεσης της οικονομικής ε, ολοκλήρωσης. Οπότε εγώ το βλέπω μόνο από την πλευρά των καταναλωτών, καταθετών, αποταμιευτών οι οποίοι μπορούν να τοποθετούν με πιο υγιή τρόπο τις αποταμιεύσεις του σε μια πιο ολοκληρωμένη αγορά. Ευχαριστούμε πολύ με αυτή την τελευταία ερώτηση. Ολοκληρώθηκε η ακρόση αυτή του Πέτρου Ματσάδο. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ξέχασα να σας ρωτήσω αν θέλετε δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε την ακρόασή σας. Όχι απλώς να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις και να σας πω ότι σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστούμε. Έχουμε πολλές ακροάσεις βλέπετε σήμερα. Ένα λεπτό διακοπή και θα συνεχίσουμε με το επόμενο. Ωραία, περνάμε στην επόμενη ακρόαση για τον ορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξηγένσης. Αυτή τη φορά έχουμε τον Χεσούς Σαντίνα που προτείνεται για μέλος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξηγένσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ακρόασή μας απορρέει από το άρθρο 56 του κανονισμού του Ενιαίου Συμβουλίου Εξηγένσης που λέει ότι το Συμβούλιο ορίζει μετά από έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τις πρακτικές που έχουμε συμφωνήσει, θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Εισαγωγικέ παρατηρήσει από τον Χεσού είναι για 5 λεπτά και στη συνέχεια 4 λεπτά ερωτήσει και απαντήσει με τη δυνατότητα συμπληρωματική ερώτηση εφόσον το επιτρέπει ο χρόνο. Κάθε πολιτική ομάδα έχει ένα χρόνο. Ε, τεσσάρων λεπτών. Εάν το επιτρέπει ο χρόνος, θα έχουμε και άλλα δύο λεπτά στη συνέχεια στη διαδικασία του Catch the Eye, σύμφωνα με ε, την στάθμιση των πολιτικών ομάδων. Και εφόσον το επιθυμεί, ο κύριος Σωρίνα μπορεί στο τέλος να κλείσει με άλλα δύο λεπτά παρέμβαση. Συνεπώς, παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Σωρίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα σε μια επιτροπή η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να προστατεύει την οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Η επιτροπή σα βοήθησε να δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση, όπω επίση και το ενίο Συμβουλίο εξηγένση Έτσι, οι Ευρωπαίοι πολίτε και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι προστατεύονται καλύτερα από τα προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο. Πέρα από έναν ευρωπαϊκό θεσμό, το νέο Συμβούλιο Εξυγίανση έχει επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Είναι μια αξιόπιστη αρχή που βοηθάει με σχέδια και με καθορισμό απαιτήσεων όσον αφορά τις σημαντικές τράπεζες στην Ευρώπη. Επίσης, επιτυχώς έχει πετύχει και την πρώτη εξυγίανση μιας μεγάλης ε, συστημικής τράπεζας της Ισπανίας το 2017. Τώρα πρόκειται για τον διορισμό μου, κάτι το οποίο με εμπνέει πραγματικά και αποτελεί για μένα μια μεγάλη πρόκληση. Συμφωνώ απόλυτα με την αποστολή του Ενίου Συμβουλίου που είναι να δημιουργεί ε, τι προποθέσει για συντεταγμένη διαδικασία εκαθάριση των τραπεζών ή εξηγένση των τραπεζών, εφόσον αυτό αποφασίζεται. Και αποτελεί ένα βασικό πυλώνα για την σταθερότητα την οικονομική στην Ευρώπη. Και έτσι μπορεί να προστατεύσει και τα συμφέροντα του κοινού. Σε όλη μου τη σταδιοδρομία, πάντα στο δημόσιο τομέα, προσπαθούσα να πετύχω αυτόν ακριβώς το στόχο. Τώρα, τι μπορώ να συνεισφέρω στον ενιαίο, στο ενιαίο Συμβούλιο Εξηγένσης. Πρώτα απ' όλα, η κατάρτισή μου. Μετά από πέντε χρόνια εκπαίδευση στα οικονομικά, και την οικονομία, απέκτησα και PhD στην οικονομία. Έπειτα, έχω και επαγγελματική εμπειρία πάνω από 25 χρόνια, οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ισπανίας σε διάφορους τομείς πραγματογνωμοσύνης που έχουν να κάνουν με τα εδώ Εξηγήση, οικονομικοί κανόνες, εποπτεία, σταθερότητα. Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ως επόπτης και μετά προχώρησα στον τομέα της ε, σταθερότητας, οικονομική σταθερότητα και μετά συνεργάστηκα και με θέματα που έχουν να κάνουν με τον κανονισμό σταθερότητας. Στη συνέχεια ασχολήθηκα με την εξυγένση ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Banco de España και ήμουνα υπεύθυνο για τα σχέδια εξυγένσης των Ισπανικών Τραπεζών σε συνεργασία με το Νέο Συμβούλιο Εξυγένσης. Στη συνέχεια ε, προσέφερα και την εμπειρία μου ως διαχειριστής 220 ατόμων από διάφορα τμήματα. Είχα την ικανότητα δηλαδή να ηγηθώ ομάδων και αποτελεσματικά μάλιστα και ιδιαίτερα πρόσκεισα και το θέμα της ε, ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Τέλος έχω εμπειρία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο που πιστεύω ότι αποτελεί ένα κόμμα προσόν για τον διορισμό μου. Τα τελευταία χρόνια ε, από την Τράπεζα της Ισπανίας συνεργάστηκα με διάφορα διεθνή φόρα, με την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το Συμβούλιο Εποπτών ε, της Τράπεζας αυτής και με το Συμβούλιο Εξηγένσης. Επιτρέψτε μου εδώ να υπογραμμίσω και κάποια επιπλέον στοιχεία της σταδιοδρομίας μου. Ήμουν υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή των όσων προβλέπονταν στην Ισπανία το 2000 2005. Ο μηχανισμός αυτός οδήγησε στη συνέχεια να φτιάξουμε το προστατευτικό σκέλος για τις τράπεζες. Κάτι το οποίο δείχνει ότι μπορώ να αναπτύξω και να πετύχω στατικικούς στόχους, αλλά και το ότι είμαι ανεξάρτητος από τον ιδιωτικό τραπεζικό κλάδο. Το αναλυτικό μου έργο επίσης υλοποιήθηκε με 25 άρθρα, τα οποία έχω δημοσιεύσει σε ε, διεθνείς εκδόσεις. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, για δύο χρόνια Έχω συνεργαστεί με το Συμβούλιο Εξυγένσης ως υπεύθυνο για την ε, ε, αποφυγή εξυγένσης στην Ισπανία. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Η εκαθάριση, η εξυγίανση, η εναρμόνιση των ε, προϋποθέσεων για την εκαθάριση, την εκαθάριση μικρών και μεσαίων τραπεζών, την αναλογικότητα και όλα αυτά για το συμφέρον των διαφερομένων. Μετά από τη μακρά μου σταζιοδρομία στην Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, το θέμα της ρύθμισης των τραπεζών, η εποπτεία αλλά και η εξυγίανση είναι πράγματα πάνω στο οποίο έχω εργαστεί και αισθάνομαι έτοιμο τώρα να δραστηριοποιηθώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο πάντα ονειρευόμουν. Εφόσον επιλεγώ για την θέση αυτή, θα χρησιμοποιήσω όλη μου την ενέργεια και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσω όλε αυτέ τι προκλήσει. Προσλέπω σε συνεργασία μαζί σα για να ενισχύσουμε την οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη, που είναι ο οίκος όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε την πρώτη ερώτηση από τον Μάρκους Φέρμπερ Ελκ. Ευχαριστώ και καλώς όρισατε κύριε Σαωρινά. Από τότε που φτιάξαμε την Τραπεζική Ένωση είχαν προβλήματα διάφορες ε, τράπεζες και τίθε το ερώτημα, φυσικά και το ερώτημα τι έπρεπε να κάνουμε με αυτές τις τράπεζες, ειδικότερα όσον αφορά το σύστημα εξυγίανση. Ε, συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις ε, έδωσαν την περίπτωση ότι η αντιμετώπιση ορισμένων τέτοιων υποθέσεων ερχόταν σε αντίθεση με το πνεύμα του μηχανισμού εξυγένση. Τι απολογισμό κάνετε εσεί αυτού του μηχανισμού εξυγένση τα τελευταία χρόνια, ποια διδάγματα αποκομίζετε από τα όσα συνέβησαν και από πλευράς αρχής, ε, τι θα βελτιώνατε, όπως επίση και στο νομοθετικό πλαίσιο. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των όσων έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Εξηγήνησης για κάποιες υποθέσεις από αυτά το οποίο έχει κάνει για άλλες. Δηλαδή, για να αποφασίσει είτε καθάριση είτε εξυγίανση, θα πρέπει να της κοινοποιηθεί τράπεζα η οποία είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας στα πέντε χρόνια που είμαστε στη θέση μας έχουμε λάβει πέντε τέτοιες υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν το Banco Popular. Θεωρήθηκε πως υπάρχει δημόσιο συμφέρον στην περίπτωση αυτή και λύθηκε με επιτυχία. Οι άλλες ε, και εξηγιάνθηκε με επιτυχία. Οι άλλες τέσσερις υποθέσεις τις οποίες αντιμετωπίσαμε είναι δύο λετωνικές τράπεζες, σχετικά μικρές και δύο ιταλικές εάν δεν λαθεύω. Εκεί δεν προχωρήσαμε σε εξυγίανση γιατί δεν θεωρήσαμε πως υπάρχει δημόσιο συμφέρον και ούτε κρίσιμες δραστηριότητες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ε, προστατευτεί. Οπότε στην περίπτωση αυτή θεωρήσαμε πως η καλύτερη λύση είναι η εκαθάριση. Υπάρχουν κάποια διδάγματα που πρέπει να πάρουμε από τις επιτυχής υποθέσεις, οπότε μπορεί κανείς να εξηγιάνει, αυτό είναι δεδομένο, τράπεζες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις περιπτώσεις που δεν προχωρήσαμε σε εξηγίανση και δεν κρίθηκε πως υπάρχει δημόσιο συμφέρον, το δίδαγμα είναι πως μπορεί τελικά να καταλήξει κανείς σε διαφορετικούς τύπους εκαθάρισης και το σενάριο που θα ακολουθηθεί θα εξαρτηθεί από τις χώρες που καλύπτεις. Δηλαδή, μπορεί να έχεις 19 διαφορετικά καθεστώτα εκαθάρισης και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το προσέξει ιδιαίτερα γιατί, για παράδειγμα, πιστωτές οι οποίοι μετά την εκαθάριση βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση γιατί η μεταχείριση που έλαβαν είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκανε. Δηλαδή είχαμε τις λετωνικές τράπεζες με δύο διαφορετικές εκαθαρίσεις ή έχουμε και περιπτώσεις όπου έχουμε άλλα εργαλεία και αυτά όταν χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της εκαθάρισης όπως έκαναν οι Ιταλικές αρχές το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Τι γίνεται με αυτό το διπλό σύστημα όπου έχει κανείς καταρχήν κοινή ε, εξυγίανση αλλά διαφορετικό καθεστώς, 19 διαφορετικά καθεστώτα εκαθάρισης. Ίσως και η εκαθάριση και τα διάφορα καθεστώτα θα πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε να είναι παρόμοια. Δεν είναι εύκολο αυτό, είναι μία από τις προκλήσεις αλλά η κατάσταση σήμερα επίσης δεν είναι ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ από τους ελιστές. Νομίζω πως ο συνάδελφος Μάρκους έθεσε σωστά τη συζήτηση για το τι πρέπει να αναθεωρήσουμε στο τρέχον πλαίσιο ε, εξυγίανσης με τα παραδείγματα που έχουμε λάβει με κάποιες τραπεζικές ε, ε, οντότητες οι οποίες χρειάστηκε να τις αντιμετωπίσουμε με διαφορετικά συστήματα τα οποία είναι στη διακριτική ευχάρεια των εθνικών αρχών όλα ήταν νόμιμα αλλά και λίγο διαφορετικά μεταξύ τους οπότε στις περιπτώσεις που εφαρμόσατε την εξυγίανση ε, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, όπως στον Banco Popular. Ποιο ήταν το δίδαγμα, μπορείτε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Σίγουρα μάθαμε κάποια πράγματα από την εξυγίανση της ε, Banco Popular Español. Το πρώτο βασικό μάθημα είναι ότι ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξηγένση τραπεζών στην Ευρώπη. Υπάρχει δυνατότητα εξυγίανσης μιας μεγάλης συστημικής τράπεζας εγχώριας ε, με συνολικό ενεργητικό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, όχι μόνο σε ένα Σαββατοκυριακό, αλλά και σε μια νύχτα. Η υπόθεση αυτή είναι σημαντική διότι δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει, να επιτύχει όλου του στόχου τη εξυγέννηση επιτυχώ. Ε, εδώ προστατεύσαμε τις κρίσιμες λειτουργίες. Με απλά λόγια σημαίνει ότι η τράπεζα άνοιξε την επόμενη μέρα τις πόρτες της. Την επόμενη, συγγνώμη, Τετάρτη το πρωί. Χωρίς ε, να προκληθεί οικονομική αστάθεια και το σημαντικότερο με απόλυτη προστασία των φορολογουμένων. Κανένα ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε ε, σε αυτή την εξυγίανση ευρώ που να προέρχεται από φορολογουμένη. Και αυτό μα δείχνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μοντέλο από το bailout που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν σε bail-in. Ε, γι' αυτό ήταν σημαντική αυτή η υπόθεση εξυγένσης. Και αυτό είναι το πρώτο δίδαγμα. Υπάρχουν και άλλα. Ένα άλλο σημαντικό είναι η συνεργασία και πόσο σημαντική είναι ε, η συνεργασία μεταξύ του SSM του SRB, των Εθνικών Αρχών Εξυγένσης και των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών. Ε, η στενή συνεργασία ήταν ιδιαίτερα εντατική και στενή μεταξύ όλων αυτών των αρχών. Το τρίτο δίδαγμα είναι ότι πρέπει να, να είναι κανείς έτοιμος ε, για ε, εξυγίανση. Δηλαδή, οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, να, κάνουν, να εξετάζουν δοκιμαστικά σενάρια, να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης, να υπάρχει ένα εγχειρίδιο για την ετοιμότητα, για αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και οι τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες για εξυγένση. Και το κλειδί εδώ είναι να υπάρχουν εικονικά, εικονικές αίθουσες δεδομένων όπου να μπορεί να γίνεται γρήγορα μια αποτίμηση, μια αξιολόγηση γιατί συχνά σε περίπτωση εξυγένσης δεν υπάρχει πολλής χρόνος για να γενικά τέτοιο. Οπότε αυτέ οι εικονικέ αίθουσε αξιολόγηση καλό θα ήταν να υπάρχουν ώστε να αξιολογούνται οι τράπεζε, να εξετάζονται διάφορα σενάρια, διάφορε διαδικασίε, ανάλυση διαφόρων πιθανών αγοραστών, ανάλυση τη κατάσταση τη τράπεζα. Πράγματα δηλαδή που μπορούν να προσταθούν στην τράπεζα από πλευρά των αρχών και από πλευρά ε, των τραπεζών. Ε, θα ήταν πολύ σημαντικά σημαντικές τέτοιες διαδικασίες και κάτι τελευταίο ε, ζητήματα που εκκρεμούν είναι η ρευστότητα σε περίπτωση εξυγένσης. Ακόμα δεν έχει πληθεί πλήρως. Στην περίπτωση της Banco Popular υπήρχε ένας πολύ μεγαλύτερος αγοραστής που ήταν έτοιμος να καλύψει το κενό ρευστότητας. Τι θα συνέβαινε όμως σε περίπτωση bail-in μιας τράπεζας που έχει εξαντλήσει όλες τις διασφαλίσεις, όλες τις εγγύησεις. Την επόμενη μέρα ανοίγει στην τράπεζα και η τράπεζα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί χωρίς ε, ρευστό διαθέσιμο. Οπότε και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο. Ε, απλά η κεντρική τράπεζα πρέπει να παρέχει τη ρευστότητα με κάποιες εγγύσεις τις οποίες ε, θα παρέχει ε, το SRF πιθανότατα. Αυτά είναι τα διδάγματα που θεωρώ ότι αποκομίζουμε από αυτό το επιτυχή εξυγένση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ερνέστε Ορτασούν από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Πρώτον, να σας ρωτήσω για την έννοια του συμφέροντος του δημοσίου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ανάλογα πως ερμηνεύει κανείς αυτό τον όρο, καταλήγει και σε διαφορετικά συμπεράσματα. Μπορεί να υπάρχει ένα ενίο πλαίσιο που να βοηθήσει με τα κριτήρια. Δεύτερον, όσον αφορά τους ε, πιστωτές, τι γίνεται με αυτούς. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν σε διάφορες εξηγιάνσεις. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Το θέμα του δημοσίου συμφέροντος και πώς αυτό αξιολογείται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δημοσιεύσει την πολιτική την οποία εφαρμόζει. Αν ε, έχει πολύ σημαντικές ε, λειτουργίες, ε, Ίσως είναι κάπως νωρίς να πούμε ότι χρειαζόμαστε επιπλέον κωδικοποίηση ή να σφίξει κάπως ε, το περιεχόμενο της έννοιας αυτής του δημοσίου συμφέροντος. Προς το παρόν πέντε περιπτώσεις είχαμε, οπότε ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα για το κατά πόσο πρέπει ε, το θέμα αυτό του δημοσίου συμφέροντος να το δούμε πιο περιοριστικά ή όχι. Για τη δεύτερη ερώτησή σας, αυτή είναι πολύ βασική για την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία BRD2 αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρος και προστατεύει τους μικρής κλίμακας επενδυτές με τις δοκιμές επιλεξιμότητας και καταλληλότητας που υπάρχουν. Ότι δεν μπορούν να επενδύσουν πάνω από 10% για παράδειγμα των ε, holdings τους σε επικίνδυνα κατά κάποιο τρόπο προγράμματα. Υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσό. Όλα αυτά αποτελούν βήματα προς τα μπρος για να προστατεύσουμε ακριβώς αυτούς τους επενδυτές μικρής κλίμακας. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω όμως ότι το ενίο Συμβούλιο Εξυγένσης μπορεί επίσης να κάνει περισσότερη δουλειά από αυτού. Μπορεί να δει καλύτερα επιτόπου τις δυνατότητες που υπάρχουν, να διπλοτσεκάρει κατά πόσο τα κριτήρια εφαρμόζονται πλήρως, κατά πόσο οι δοκιμές αυτές καταλληλότητας είναι σωστές και ενδεχομένω να δούμε αν υπάρχουν εμπόδια στην εξυγίανση εφόσον όλα αυτά δεν γίνονται ικανοποιητικά. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι υπάρχει ανάγκη για μια αλλαγή νοοτροπίες στις τράπεζες και στους τραπεζικούς ομίλους για να καταλάβουμε ότι το μη selling είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται το θέμα των ακάλυπτων δηλαδή και ότι είναι κάτι το οποίο οδηγεί και σε λειτουργικούς κινδύνους στις τράπεζες. Άρα και προβλήματα με τέτοια κεφάλαια. Ευχαριστώ, πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με τον κατάλογο των ομιλητών που βρίσκονται στην αίθουσα. Θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις ή κάποια σχόλια. Σας ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, αξιότιμοι Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο στο να με ακούσατε και σας ευχαριστώ για τις παραπάνω που ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Ήταν τιμή που ήρθα να με ακροαστείτε εδώ, ε, σε αυτή την επιτροπή που βοήθησε τόσο πολύ στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Σας ε, λέω πως για το θέμα αυτό θα εργαστώ με όλη την εμπειρία που έχω, που είναι επαρκής και ε, θα έπρεπε να γίνω ε, ε, πλήρες μέλος του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης προσφέροντας τις επαγγελματικέ μου γνώσεις και πάντα με πνεύμα συνεργασίας για να διδαχτώ από τους συναδέλφους και να πετύχω τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα των Ευρωπαίο πολίτη. Εάν με διορίσετε να ξέρετε πως θα είμαι πάντα ανεξάρτητος και δεσμεύομαι πως θα προωθήσω το δημόσιο συμφέρον λογοδοτώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάντα θα είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ μαζί σας για να βελτιώσουμε ε, τις διαδικασίες εξυγίανσης και οικονομική σταθερότητα σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ μερικά λεπτά διάλειμμα πριν περάσουμε στην επόμενη ακρόαση.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 with each other. So they needed a new uh, chair. Okay. I think... Καλησπέρα σας. <laughs> I think we can... Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε με την τρίτη ακρόαση που θα κάνουμε σήμερα το απόγευμα. Είναι ο διορισμός του Αντιπροέδρου ε, του Ενίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, καλωσορίσω, κύριε Ζωάντε Καρπενθιέ. Σας έχουν προτείνει ως υποψήφιο για την Αντιπροεδρία για τη θέση αυτή και πρέπει να σας πω ότι εδώ είμαστε ευθυγραμμισμένοι με το άρθρο 56 του κανονισμού για το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης που ορίζει πως το Συμβούλιο εγκρίνει μία εφαρμοστική απόφαση για τον διορισμό της Προεδρίας, Αντιπροεδρίας και των τεσσάρων μελών με πλήρη δικαιώματα σύμφωνα από την έγκριση με, ε, δόντας την έγκριση της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με εισαγωγικά ε, σχόλια, 5 λεπτά, μετά 4 λεπτά ερωτήσεων και απαντήσεων με σλότ για τις συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες και αν το επιτρέψει ο χρόνος θα έχουμε και επιπλέον σλότ των 2 λεπτών σύμφωνα με τη διαδικασία Catch the Eye λαμβάνοντας υπόψη ε, και του βάρους των πολιτικών ομάδων. Και αν το επιτρέπει ο χρόνος και το επιθυμεί, θα καλέσω τον κύριο Καρπετιέ να κάνει και κάποιες καταλεκτικές παρατηρήσεις, μετά ε, οι οποίες θα φτάνουν μέχρι τα δύο λεπτά. Σας δίνω το λόγο λοιπόν κύριε Ντεκαρπεντιέ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα. Και μιλώντας για το θέμα της εξυγίανσης των τραπεζών στην Ευρώπη και το σχετικό συμβούλιο είναι να μιλά κανείς για ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες γιατί το να μπορεί κανείς να εξυγείανει και να εκαθαρίζει μια τράπεζα έχει να κάνει με τις με τις ε, ανάγκες που έχουμε να εξασφαλίσουμε το τραπεζικό σύστημα ε, σήμερα και στο μέλλον. Όταν με ρωτάνε τα παιδιά μου τι κάνω, καταρχήν πρέπει να τους εξηγήσω και δυσκολεύομαι γιατί χρειάζεται και πόσο σημαντικό είναι για την καθημερινότητα. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι οι βασικές εμπειρίες που απέκτησα κατά τη διάρκεια της επαγγελματική μου σταδιοδρομία, για παράδειγμα, κατέρευση των Ισλανδικών τραπεζών το 2006 που δημιούργησαν τεράστιε κοινωνικέ εντάσει και προβλήματα ε, στην Ισλανδία. Πήρα ταξί από το αεροδρόμιο στο Ρέικιαβικ ε, και στη μισή ώρα που ε, ήμουν στο ταξί μου, είπε ο ταξιτζής πω έχασε την επιχείρηση και δούλευε ω ταξιτζής, έβαλε το σπίτι του να πουληθεί και δεν ήταν μόνο ο οικονομικό αντίκτυπο στον οποίο αναφέρθηκε, αλλά και στην διαταραχή τη προσωπική του ζωή, τη καθημερινή ζωή, ζωής, της οικογενειακής τη ζωής, της ζωή τη κοινότητά του. Άρα λοιπόν είναι παραπάνω από επάγγελμα για μένα ο, το ενιαίο Συμβούλιο εξυγίανση. Είναι ένα τρόπο για να σταθεροποιήσουμε την Ευρώπη και έχουμε ένα κεντρικό ρόλο ε, στην εξυγίανση της ε, χρηματοπιστωτικής εικόνας στην Ευρώπη. Όλο και περισσότερο έχουμε κάνει σε αυτά τα τέσσερα χρόνια στα οποία εργάζομαι εκεί και είναι πολλές οι προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται. Δηλαδή θα πρέπει να είναι φερέγγες οι τράπεζες υπό όλες τις συνθήκες και αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό μεμονωμένα στο ενιαίο Συμβούλιο Εξυγένσης αλλά σε στενή συνεργασία με τον τραπη... με τραπεζικό ε, ε, κύκλο με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης όπως επίσης και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα χρειάζεται τα δικά μας, ε, οι δικές μας αρμοδιότητες, οι οποίες είναι παρεμβατικές, να εξισορροπηθούν από τη λογοδοσία και τη μέγιστη διαφάνεια. Και πιστεύω πως με την ομάδα μου το έχουμε καταφέρει κάθε μέρα υπό δύσκολες συνθήκες. Και φιλοδοξία μου είναι να διατηρήσουμε τη συνεισφορά μας στην πλήρη εφαρμογή του ε, πλαισίου για την εξυγίανση υπό τον τρέχοντα ρόλο και είμαι έτοιμος και θα αναλάβω και περισσότερες αρμοδιότητες εάν διοριστώ ως αντιπρόεδρος του Ενίου Συμβουλίου Εξυγίανσης γιατί έχω ε, ε, από την χρηματοπιστική εποπτεία και από τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων αρκετή εμπειρία για να μπορώ να συνεισφέρω στη μεγαλύτερη επιτυχία του Συμβουλίου Εξυγένσης στο μέλλον. Και τέσσερα είναι τα σημεία στα οποία θα τονίσω, δηλαδή επικοινωνία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα ε, της κρίσης των αρμοδιοτήτων ε, και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δεκαρπέντιε. Πάμε στις ερωτήσεις και ξεκινάμε τον Μαρκούς Φέρμπερ του ΕΛΚ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντεκαρπεντιέ, καλώς ορίσατε. Αν δεν σας πειράζει να μιλήσω γερμανικά. Το 2019 το Νοέμβριο το δικαστήριο έλαβε τρεις αποφάσεις ε, για εξάντε ε, τέλη για την Banco Cooperativa Español και για άλλες δύο τράπεζες. Και, τα, και δήλωσε ότι αυτά τα τέλη ήταν ε, παράνομα. Η απόφαση αυτή να δηλωθούν τα τέλη ε, άκυρα βασίστηκαν στην επέκταση του Single Resolution Fund ε, μικρά λάθη μπορεί να οδηγήσουν ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη και πώς ε, τι θα γίνει με τέτοιες αποφάσεις που θα ληφθούν στο μέλλον Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντική απόφαση του, του δικαστηρίου. Το δικαστήριο αυτό έλαβε αυτές τις αποφάσεις για τρεις τράπεζες ε, για εξάντε ε, τέλη και αυτό βασιζόταν σε διαδικαστικά προβλήματα. Για να σας εξηγήσω το υποβαθρό και έχετε δίκιο. Ε, το Γενικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίξει τη θέση ε, του SRB το 2016 η έμφαση ήταν στο να γίνουν σωστά οι υπολογισμοί. Ήταν ένα περίπλοκο σύστημα το οποίο απαιτούσε ε, ερμηνεία από τη νομική υπηρεσία και δόθηκε έμφαση στο να γίνει σωστά υπολογισμός. Ταυτόχρονα όμως όπως αποφάσισε το δικαστήριο διαδικαστικά τα πράγματα δεν έγιναν όπως έπρεπε. Οπότε τελικά αποφάσισε να ακυρώσει το δικαστήριο αυτές τις τρεις αποφάσεις Γεγονό που σημαίνει ότι η Σερβία πρέπει να λάβει νέε αποφάσει για αυτέ τι ε, τράπεζε να αποσύρει την νομική βάση και να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια θα έμεναν εκεί που έπρεπε στο SRF. Δηλαδή, ε, πράγματι υπήρξαν προβλήματα και θα ήθελα να αποφύγουμε φυσικά τέτοιε ε, ελλείψεις διαδικαστικέ, αλλά από την αρχή η έμφαση ήταν στο να γίνει σωστό υπολογισμό, Αλλά από νομική άποψη διαπιστώθηκε ότι διαδικαστικά ήταν το πρόβλημα που δημιούργησε πρόβλημα στις τράπεζες ώστε τα κονδύλια τελικά έμειναν στο SRF εκεί που έπρεπε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, ναι. Στην προετοιμασία τις απόφασεις του δικαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί ώστε να αποφευθούν τέτοια λάθη στο μέλλον. Δηλαδή το Ταμείο εξηγένση, ε, θα μπορούσε να μεγαλώσει όπω έχει σχεδιαστεί. Ναι, σίγουρα. Πρέπει να αποφεύγουμε τέτοια σφάλματα ε, και τα διαδικαστικά προβλήματα. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω, ωστόσο, ίσω να μην ήμουν απόλυτα σαφή, είναι ότι ο λόγο που ακυρώθηκαν οι τρει αποφάσει σχετικά με τι τρει τράπεζε για σχετικά μικρά ποσά ήταν διαδικαστικός ώστε να αποκατασταθεί η νομική βάση και να ληφθεί μια νέα απόφαση για τις τρεις τράπεζες για να αποκατασταθεί η νομική βάση ώστε να μείνουν τα κονδύλια εκεί που ήταν. Όπως το βλέπω εγώ, δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπήρχε λόγος τελικά να καταβάλει αυτά τα τέλη τράπεζα για το 16 αυτές τις τράπεζες οπότε έτσι ακυρωθήκε η απόφαση ευχαριστούμε πολύ Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια εργαστήκατε στον, στο Συμβούλιο αυτό και θέλω να μου μιλήσετε λίγο για την εξηγίαση της Banco Popular και τα νομικά προβλήματα τα οποία συνδέθηκαν με την απόφαση αυτή εξηγίανσης της τράπεζας όπως επίσης θέλω να μου πείτε και για τα θέματα διαφάνειας μετά από την απόφαση όσον αφορά τις δυσκολίες δηλαδή ε, τις επιπλέον ε, πληροφορίες που δικαιολογούσαν την εξυγένση. Υπήρξαν προβλήματα διαφάνειας, διαφάνειας που συνδέονται και με νομικά ζητήματα. Οπότε κατάλαβα, εσείς ήσασταν στο νομικό τμήμα του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης. Οπότε μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για την εξυγένση αυτή τη συγκεκριμένη τράπεζα. Ευχαριστώ. Μετά την απόφαση εξυγένσης για την Banco Popular υπήρξε ένας μηχανισμός πρόσβασης στα έγγραφα. Τότε η αξιολόγηση έγινε με τη δέωση επιμέλεια δόθηκαν οι πληροφορίες. Όμως, αυτοί που προσβλήθηκαν από την απόφαση ε, προσέφυγαν και ζήτησαν περισσότερη διαφάνεια. Και αυτό που κάναμε εμείς και το συζητήσαμε μήνες μετά από την απόφαση για την εξηγένση, δόθηκαν επιπλέον πληροφορίες. Όταν λήφθη η πρώτη απόφαση για την διαφάνεια, κάναμε μία αξιολόγηση του νομικού πλαισίου και των διαφόρων συμφερόντων. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα της διαφάνειας, υπάρχει και η οικονομική σταθερότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη και άλλοι παράγοντες. Οπότε νομίζω ότι η προσέγγιση μας δικαιολογόταν. Αλλά ο κόσμος ζητάει περισσότερη διαφάνεια και αυτό προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε αμέσως. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν νομικά κολλήματα όσον αφορά τις ε, νομικές διαδικασίες. Η απόφαση για περισσότερη διαφάνεια τέθηκε σε εφαρμογή αμέσως. Και ακολούθησαμε αυτή τη διαφάνεια και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Αν ήμασταν, είχαμε περισσότερη διαφάνεια από την αρχή, είναι δύσκολο να πει κανείς αν θα ήταν καλύτερη κατάσταση ή όχι τώρα εκ των υστέρων. Πρέπει να ζυγίσουμε πολύ καλά τα διάφορα συμφέροντα ανά πάσα στιγμή. Η προσέγγιση μας νομίζω ότι ήταν καλή. Μερικούς μήνες αργότερα η εξολόγηση ήταν διαφορετική και χρειαζόταν περισσότερη διαφάνεια, την οποία και δώσαμε τότε αμέσως. Ευχαριστούμε Λουίς Καρικάνο. Ρινιού. Συγγνώμη, συγγνώμη στο Ολλανδικά, ο κύριος Γκαρικάνο, έχασα την παρουσίασή σας στην αρχή και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας για το κατάλληλο επίπεδο παρέμβασης από πλευράς του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Είναι σωστό που έχει τέτοιο υποπτικό ρόλο το Συμβούλιο αυτό και που αποφασίζει στην πράξη να αποφασίζει για το θέμα του κοινού Ε, πρόκειται να επεκταθεί και νομικά ο ρόλος του Συμβουλίου. Για να το πω πιο ξεκάθαρα, θα αναγκαστεί να λαμβάνει δράση το Συμβούλιο. μήπως θα έπρεπε να αλλάξει κάπως το θέμα του κοινού συμφέροντος και να ε, μπορεί να προχωρήσει σε εξυγίανση αντί για εκαθάριση, να είναι αυτός ο κανόνας. Υπάρχει βέβαια η οδηγία BRD φυσικά που καθορίζει κάποια κριτήρια. Τώρα ξέρω θα μου πείτε ότι θα θέλατε εναρμόνιση στην εκαθάριση. Εντάξει, αλλά δεν μου φτάνει εμένα αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι η εναρμόνιση στην εκαθάριση είναι κάτι το οποίο θα δούμε ε, κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Ίσως ε, θα έπρεπε το Ενίο Συμβούλιο να βρει άλλους τρόπους για να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση Αν ο κανόνας εξεκολουθεί να είναι η καθάριση και αν ε, οι χώρες πρέπει να διασώσουν τις τράπεζές τους, ε, εάν γίνει αυτό με κάποια τράπεζα θα πάμε πίσω σε αυτά που είδαμε την ε, προηγούμενη δεκαετία. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσα ρωτήσατε. Αν εξετάσει κανείς τι ε, τις αποφάσεις μας, η πρώτη ήταν μια εξυγίανση και έπρεπε να αποφασίσουμε ότι αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον. Και όχι, δεν υπήρχε, άρα λοιπόν πέρασαν από την εθνική διαδικασία καθάρισης. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα του τρέχοντας πλαισίου που δίνει ένα κατόφλι ξεκάθαρο και λέει ναι ή όχι. Άρα λοιπόν η, η βασική εναλλακτική, εάν δεν προχωρήσουμε σε εξηγήνση, είναι η καθάριση. Σε εθνικό επίπεδο τώρα, κατά πόσο θα ε, διευρύνουμε το πεδίο και θα το επεκτείνουμε, είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσω εγώ αυτό. Ίσως ε, μπορεί να ε, ε, διευκρινίσουμε καλύτερα και να ορίσουμε τι σημαίνει δημόσιο συμφέρον ή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ποια περίπτωση εκαθαρίζεται, σε ποια περίπτωση εξηγένονται οι τράπεζε. Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο να το περιγράψει κανεί παρά να το κάνει. Και το τρέχον πλαίσιο δίνει μια ισορροπημένη προσέγγιση. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να προδικάσει κανεί το μέλλον και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, Υπάρχει λόγος να εξηγιάνουμε άλλη τράπεζα. Ή θα στείλουμε άλλες τράπεζες σε εθνική εκαθάριση. Θα διευρυνθεί ο ρόλος μας, θα επεκταθεί. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να σας απαντήσω. Έχετε όμως δίκιο. Θα πρέπει ο νομοθέτης ενδεχομένως να αλλάξει το κομμάτι που αναφέρεται στο δημόσιο συμφέρον. Έτσι χαμηλώνει ο πύχης και είναι πιο εύκολο να περάσει κανείς σε εξυγίανση. Και τότε στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο θα συμμετέχει πιο πολύ και δεν θα βασίζεται τόσο στα πτωχευτικά συστήματα κάθε χώρας. Είναι ένα ισορροπημένο πλαίσιο, αυτό πιστεύω, και θα κατέληγα στο εξή. Παρόλο που ε, είχαμε κάποιες αρνητικές αποφάσεις, δηλαδή όχι εξυγίανση αλλά η καθάριση σε εθνικό επίπεδο, αυτό δεν μπορεί να προδικάζει το μέλλον. Τώρα, είμαι πιο αισιόδοξο από ότι είστε ε, Βέβαια είστε σε καλύτερη θέση από μένα να γνωρίζετε τι θα γίνει με το θέμα το δεύτερο, αλλά ελπίζω προσωπικά πω οι εξελίξει θα είναι θετικέ και θα εναρμονιστούν τα εθνικά πτωχευτικά συστήματα και θα υπάρχει ένα ενιαίο ε, σύστημα ε, εκαθάρισης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ο κύριος Ουρτασούν, εκ μέρους των Πρασίνων, ευχαριστώ πολύ. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ως αντιπρόεδρος θα είστε ε, υπεύθυνο για το Ταμείο. Οπότε, οι βασικές αποφάσεις για την ακύρωση ε, τριών εκ των προτέρων συνεισφορών το 16 σε τι διδάγματα μας οδήγησαν. Και για τον Banco Popular, το Δεκέμβριο φέτος, ελήφθη μία απόφαση για την αποζημίωση ή όχι ε, όσους είχαν ομόλογα ή μετοχές της τράπεζας αυτής. Και η απόφαση αυτή αν... αναβλήθηκε και πάλι ε, περίεργο γιατί εξηγιάνθηκε το 2017 ή μέσα στο 2020. Γιατί καθυστερεί αυτή η απόφαση γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ε, κομμάτι των αρμοδιοτήτων σας, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν αυτές τις αποφάσεις του 2016 του δικαστηρίου που ακύρωσε τον υπολογισμό, μάλλον όχι τον υπολογισμό αλλά την απόφαση για τρεις τράπεζες Δηλαδή χρειάζεται να ληφθεί νέα απόφαση η οποία να βασίζεται ε, σε κάποια άλλη βάση γιατί διαδικαστικά ήταν προβληματική δείχνει πόσο σημαντικό είναι οι αποφάσει να λαμβάνονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Εν τω μεταξύ, έχουμε ε, ενισχύσει τη γραμματεία μας έτσι ώστε όλα τα διαδικαστικά κομμάτια στη λήψη αποφάσεων να εφαρμόζονται σωστά η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη στην αρχή όταν ξεκινήσαμε και όπως σας είπα σε νομικό επίπεδο προσπαθούσαμε να ε, έχουμε κάνει σωστά τον υπολογισμό χωρίς όμως να εξασφαλίζουμε πλήρως τη νομική βάση και γι' αυτό το δικαστήριο κατέληξε πως χρειάζεται νέα απόφαση για αυτές τις τρεις τράπεζες. Ποια είναι τα διδάγματα. Η ανάγκη για επαρκείς πόρους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεων και έτσι ώστε όλα να ακολουθούν το γράμμα του νόμου και για την περίπτωση της τράπεζας Banco Popular, αποζημίωση ή όχι, ξέρετε πως έχει γίνει μια προσωρινή αξιολόγηση και υπάρχει και το δικαίωμα της ακρόασης που έχει οδηγήσει σε ένα τεράστιο αριθμό σχολείων που θα πρέπει να διαβαστούν και να αξιολογηθούν και από εμά αλλά και από τους ε, εξωτερικούς ε, αξιολογητές. Είναι μια διαδικασία η οποία όντως έχει χρειαστεί πολύ χρόνο. Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της διαδικασίας και πριν τα τέλη της χρονιάς εκδώσαμε μία ανακοίνωση, οπότε είμαι αισιόδοξο πως κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος, θα ληφθεί η απόφαση Υπάρχει διαδικασία ε, του δικαιώματος ε, ακρόασης έτσι ώστε οι απόψεις να εκφραστούν και αφού εκφραστούν να αξιολογηθούν. Και αυτό χρειάζεται χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επισπεύσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο επιμελείς. Να δείξουμε τη δέουσα επιμέλεια για να φαίνεται ότι η διαδικασία είναι πλήρης και ουσιαστική. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε, έχετε και δύο λεπτά τώρα για τα τελικά σας ε, λόγια. Σας ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση εδώ. Ήταν μεγάλη μου τιμή που βρέθηκα εδώ στο Κοινοβούλιο σήμερα. Ελπίζω να απάντησα επαρκώς τις σημαντικές ερωτήσεις, ειδικότερα αυτές ε, που αναφέρονταν στις 60 αποφάσεις σωστός ε, τρόπο εξηγένση των τραπεζών εξυπηρετεί όλου του πολίτε και δεν μπορούμε να το επιτυγχάνουμε από μόνοι μα. Πρέπει να ενισχύουμε τη στενή συνεργασία με όλου του ενδιαφερομένου και το Κοινοβούλιο. Και εγώ φιλοδοξώ να συνεχίσω να συμβάλλω σε αυτό το σημαντικό έργο. Είμαι έτοιμο να αναλάβω περισσότερε ε, ευθύνε ω αντιπρόεδρο και σα διασφαλίζω ότι ω αντιπρόεδρο θα αναλάβω πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα και την εντολή θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμβάλλω σε αξιόπιστη διαφανή και χωρίς αποκλεισμού χρήση του μηχανισμού εξυγένσης ε, ε, ως σημαντικού πυλώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ τερματίζεται η συνεδρίαση για σήμερα το απόγευμα και θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί με την ε, κοινή συνεδρίαση με την ΕΜΒΗ στις 9 το πρωί. Ευχαριστούμε.